Δεν θα είναι εδώ ο κύριος Ντέβα σήμερα τελικά. Να θυμίσω στους συναδέλφους το είπαμε χτες ότι 11.30 θα σταματήσουμε λόγω της ειδική τελετής για τα 60 χρόνια της υπογραφής της συνθήκης της Ρώμης. Και να θυμίσω ότι στις 5.30 έχουμε κοινή συνεδρίαση με τον προϋπολογισμό και τις εξωτερικές υποθέσεις και η συνεδρίαση θα γίνει σε μια μεγαλύτερη αίθουσα. Νομίζω την, την 4Q2 ή την 2Q2 κοιτάξτε το πρόγραμμά σας. Πάντως στις 5.30 είναι το 2Q2. Πεντέμιση ώρα. Κοινή συνεδρίαση. Καλώς λοιπόν να ελέγξουμε τις κάρτες μας αν δουλεύει το σύστημα. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Όχι, δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Παρακαλώ βγάλτε τις κάρτες σας και ψηφίστε. Ελέγχουμε λοιπόν να δούμε αν πράγματι δουλεύει το σύστημα. Εντάξει, φαίνεται ότι δουλεύει. Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις για την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με, το, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εγγύησεις για εξωτερικές δράσεις. Ο κύριος Βέντε έχει ζητήσει το λόγο. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις κάρτες μας, εγώ και ο συνάδελφος, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε παρόλα αυτά. Εντάξει, όταν ε, πάρετε την κάρτα σας θα σας προσθέσουμε, λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος δεν έχει την κάρτα του, θα ξεκινήσουμε όμως. Με την 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Against κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 12 ψηφίζεται ψηφίσατε όλοι απερίφθη Δεκατρία υπέρ κατά αποχές απερίφθη δύο υπέρ κατά αποχές απερίφθη 14 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, περνάμε στη 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 18. Ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθηνη. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 19 ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τοπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η έλεγχος πάλι παρακαλώ για την 1. Τι είναι αυτό. Τέλος της ψηφοφορίας. Τοπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 10. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Λοιπόν, ονομαστική κλίση για την γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Μεγάλη πλειοψηφία. Δέκτη. Συγχαρητήρια λοιπόν στον απόντα εισηγητή. Περνάμε στο 9. Το δεύτερο τμήμα του πακέτου για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ο Δίβα λοιπόν ήταν για μια ακόμα φορά ο εισηγητής. 50-59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ κατά αποχές α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 70 ψηφίζεται τέλος απερίφθη 71 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για το 71 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελεκτρονικός έλεγχος για την 72 ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφη. 73 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 75 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη, 76 υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος για την 76 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε στις ψηφοφορίες. Δεκτή. 78 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 79 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 79 ψηφίζεται τέλος δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 80 Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απερίφθη. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί εγώ βλέπω διαφορετικά πράγματα. Τέλος. Δεκτή. 82 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 82. Τέλος. Δεκτή. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 87 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 87 ψηφίζεται ψηφίσατε όλοι τέλος δεκτή συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος για την 91 Τέλος. Δεκτή. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α... Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται για την 92. Τέλος. Δεκτή. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 93. Τέλος. Απερίφθη. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Για τα παραρτήματα, οι 20 και 21 ψηφίζονται από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 22 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22. Τέλος. Δεκτή. 23 και 24 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη αιτιολογικές σκέψεις 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 30 τέλος δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 9 συμβιβαστική υπέρ. Α, συγγνώμη. 5, 5. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 5. Ψηφίζεται. Κατά. Απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται τέλος δεκτή συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 50 ίδια πλειοψηφία, αλλά ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ. Κατά αποχές απερίφη. 57 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 57. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της νομοδότησης με ονομαστική κλίση. Ψηφίζετε; Τέλος. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Ντίβα για δεύτερη φορά. Να ευχαριστήσω και τη Λίλη που είναι η τελευταία ημέρα της εδώ σήμερα. Έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και επιστρέφει στην Ιταλία. και ένα συνάδελφος από τη γραμματεία που θα έρθει αργότερα φεύγει για να πάει να δουλέψει στην Άνω Βουλή. Θα τον χαιρετήσουμε αργότερα. Τώρα οι πρωτοπόρες αν θέλετε πρωτοβουλίες στον τομέα του ροχισμού. Σημαντική έκθεση και θα δώσω τον εισηγητή. Ε, η Λόλα μήπως έχει να πει κάτι πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Εντάχει θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που ε, εργάστηκαν, Σένφιλ, Ζούντιτ, και πιστεύω ότι αυτό έχει, αυτή η έκθεση έχει μεγάλη σημασία για την καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων και πιστεύω ότι θα, θα φτάσουμε στην Ολομέλεια ακόμα πιο δυνατή, διότι αυτό το θέμα μας έχει ενώσει όλους. Έχουμε έναν μακρύ κατάλογο, αλλά βλέπω ότι έγινε και μεγάλη εργασία για να φτάσουμε στους συμβιβασμούς. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και ενεκρίθη. Σελίδα 5 στο δικό μου κατάλογο. Συμβιβασμός 14. 14 υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 185 ελέγχουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 115 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-12. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές ας ελέγξουμε. 123 ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 132 άρχητη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 133 άρχιτη ψηφοφορία.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 Σελίδα 12. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 155. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 11 υπέρ. Συμβαστική. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε τη συμβαστική 12 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. 171. Νομίζω ότι εγκρίθηκε αλλά ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 174. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε τη συμβαστική 13. Έρας Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές Ελέγχουμε την 180, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 182, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 186-87 μαζί ε, υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε τις δύο αυτές τροπολογίες, 186-187, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο για τον έλεγχο. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις, μάλλον 21 υπέρ. Κατά, αποχές ελέγχουμε την 21 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 22 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 24 υπέρ κατά, αποχές, ελέγχουμε την 24, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. Ε, ε, έτσι κι αλλιώς, ε, έτσι κι αλλιώς απορρίπτεται με ή χωρίς την κάρτα σας. 23 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 23. Άρα ελέγχουμε και την κάρτα σας. Εντάξει, ωραία. Πέρας, εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε την 25 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε και την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 27 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. της 27 πέρας και εγκρίνεται. 28 και 83 από κοινού. Είναι παρόμοιες υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε 28 και 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά, αποχές, ελέγχουμε την 30. Άρχεται η ψηφοφορία, νομίζω ότι εγκρίνεται, πέρας, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 31, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι πέρας, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 36 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 56 άρχεται η ψηφοφορία νομίζω ότι απορρίπτεται πέρας ναι πράγματι απορρίπτεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε 17 πέρας ναι, νομίζω ότι με μεγάλη πλειοψηφία έχει εγκριθεί. Ακόμα και χωρίς την κάρτα σας δεν υπάρχει θέμα. Συμβαστική 18, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε την 72 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76, 77, α, όχι, καταπίπτει. 79, 79, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνε. Συμβαστική 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνε. 82, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνε. 84, που, όπου υπάρχει και μία προφορική Τη βλέπετε κάτω-κάτω. Ψηφίζουμε με την προφορική λοιπόν, εντάξει. 84 με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 1 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκλένουν, ε, ε ελέγχουμε συγγνώμη την τροπολογία 2 άρχεται πέρας και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψήφια 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 6 γιατί ψηφίζεται διαφορετικά κάθε φορά. Άρχεται η ψηφοφορία στην 6. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8. 8. Υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 8 άρχεται, η η... άρχεται ο έλεγχος πέρας εγκρίνεται τοπολογία 9 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνει. 18 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 18, άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, όχι, πέρασε, πέρασε. Είναι σαφές. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, γνωμοδότηση άλλων επιτροπών ίντα. Α. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. M υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε το M, την αιτιολογική σκέψη M. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3 της ΣΥΝΤΑ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Παράγραφος 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 ξεχωριστή ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Α, όχι, καταπίπτει. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα ελέγχουμε. Ελέγχουμε το τρίτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχατε δει και ο κύριε Βέντα ότι έπρεπε να ελέγξουμε. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, όχι, όχι, έχει περάσει. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Έχετε δίκιο. Παράγραφος 17 υπέρ κατά, αποχές, ελέγχουμε την παράγραφο 17, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. Παράγραφος 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 23, υπέρ. Α, με συγχωρείτε, ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 23, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας και απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε το τρίτο τμήμα της 23, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την Επιτροπή Απασχόλησης, αιτιολογική α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Δ, υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε το D, την αιτιολογική D. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται. Παράγραφος 3 της ΕΜΠΛ υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την παράγραφο 3, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την παράγραφο 7 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι εγώ ξέχασα να ψηφίσω γι' αυτό λείπει κάποιος εγώ ήμουν πέρας απορρίπτεται ευτυχώς που ψήφισα παράγραφος 8 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την παράγραφο 8 άρχεται η ψηφοφορία όχι, όχι, σαφώς, σαφώς απερίφθη. Παράγραφος 11 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε την 11, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την παράγραφο 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 25. Υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται, όμως ε, ελέγχουμε, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, ναι πράγματι, εγκρίθηκε. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την έκθεση στο σύνολο της όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται η έκθεση με πλειοψηφία και μερικές αποχές. Να σας συγχαρούμε για την έγκριση αυτή. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη περίπλοκη ψηφοφορία για σήμερα. Ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνάδελφοι, τι θέλετε, διάλειμμα. Δυστυχώς ε,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

Okay, colleagues, we can make a start now um, on item 11, which is... Πάμε στο σημείο υπαριθμών 11, που είναι γνωμοδότηση δημοσιονομική κανόνε που εφαρμόζονται στο Γενικό Προεπλογισμό της Ένωσης. Εγώ είμαι συντάκτρια της γνωμοδότησης. Το όλο θέμα είναι, έχει ως εξής μαζί με την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αλλάξει τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα να απλουστευτούν κάποιοι κανόνες ε, ε, βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χορηγεί κονδύλια σε εξωτερικές ομάδες. Το Φεβρουάριο είχαμε μία συνάντηση όπου ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψή και είχαμε και ανταλλαγή απόψεων με δικαιούχους ενωσιακών κονδύλιων. Ορισμένοι εξ αυτών μου υπέβαλαν τα σχόλιά τους, ε, τα οποία τα έλεγα και εγώ υπόψη μου στη γνωμοδότηση που σας καταθέτω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να περιορίσει το βάρος σε εκείνους που εκτελούν ενωσιακά προγράμματα. Και ένας ε, ένας λόγος ή ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό είναι να περιστούν έλεγχοι. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι δεχόμαστε τον έλεγχο από τον Εθνικό Οργανισμό δεν χρειάζεται να κάνουμε κι άλλον ένα. Με τον τρόπο αυτό απλουστεύονται οι διαδικασίες ε, ε, συμπεριλαμβανομένης και κάποιας θελούσιας εργασίας. Ε, νομίζω ότι και αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο θα υπάρξει ένα νέο σύστημα ανάλυσης ε, το οποίο σημαίνει, με βάση τα αποτελέσματα, που σημαίνει ότι το κονδύλι θα εξαρτάται από το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και μια άλλη μεταρρύθμιση που εισήχθη είναι ότι περιορίζεται το κόστος ε, το λογιστικό. Νομίζω ε, για τα περισσότερα από αυτά τα θέματα προτείνω να στηρίξουμε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πράγματι να καταστήσουμε απλούστερους τους κανόνες. Και όπως σας είπα, εγώ έχω κάποιες τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο να καλύψουν ε, κάποιες ε, ανησυχίες. Οι αλλαγές λοιπόν που έχω εγώ είναι οι εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ένα μαξιλάρι ευελιξία Το 10% μπορεί να ε, παρακρατηθεί στις ε, αρχές του έτους. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Ε, χρειαζόμαστε την σαφήνεια. Και εγώ έχω μια τροπολογία που λέει ότι αν αυτό το κονδύλι δεν δαπανηθεί, τότε θα πρέπει το κονδύλι να επανέλθει στο χρηματοδοτικό εργαλείο από το οποίο προήλθε. αυτό, αυτή είναι η ευελιξία. Αν έχει έρθει από ένα συγκεκριμένο προϋπολισμό θα πρέπει να επανέλθει σε αυτόν και θα πρέπει να υπάρχει μια ε, διαδικασία όπου το Κοινοβούλιο θα έχει έτσι τη γενική εικόνα του όλου θέματος. Στα στο σύστημα πληρωμών που βασίζεται στα αποτελέσματα, ορισμένοι οργανισμοί λένε δέχονται το σύστημα, αλλά πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους βασικούς κανόνες. Με ποιους θα μετριούνται τα αποτελέσματα. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει στον δημοσιονομικό κανονισμό να αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι οργανισμοί επιθυμούν να έχουν κάποια σαφήνεια πρέπει και εδώ να υπάρχει κάποια ευελιξία. Ξέρετε ότι κυρίως ε, στην ΕΚΟ, στην ανάπτυξη, ε, τα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία σε αυτό το σύστημα που θα μετράει τα αποτελέσματα. Και μια άλλη δυνατότητα είναι να δούμε πώς λειτουργούν τα καταπιστεύματα. Όπως ε, γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι είναι απαραίτητα τα καταπιστεύματα, αλλά θέλει να έχει καλύτερη υποπτία αυτών των καταπιστευμάτων. Έχουμε λοιπόν τροπολογίες που κάνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το ε, Κοινοβούλιο να μπορεί να παρακολουθεί ε, τα διοικητικά συμβούλια των καταπιστευμάτων και το δεύτερο, ε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να μπορεί να λειτουργήσει το Ταμείο, αλλιώς να υπάρχει κατεξοσεντότηση πράξη. Γιατί νομίζω ότι όλα τα καταπιστεύματα που φετρώνουν σαν τα μανιτάρια θα πρέπει κάπως και να ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτιμούμε λοιπόν όσον αφορά τις γενικές δαπάνες να υπάρχει προσαρμογή στο 7% και κατά τα άλλα αυτές είναι οι βασικές προτάσεις που καταθέτω. Η δική μας επιτροπή δεν θίγεται, θίγονται περισσότερο άλλες επιτροπές ή εξωτερικών υποθέσεων, χάρη ε, που θα επηρεαστεί πάρα πολύ από τα ε, ταμεία ε, γειτονίας. Αυτά έχω να σας προτείνω και περιμένω τα σχόλια από τους συναδέλφους μου. Δεν ξέρω αν θέλετε συνάδελφοι να πείτε κάτι. Ο κύριος Παουλ ε, Ρούμπιχ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Λίντα. Το βήμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κυρίως στην αναπτυξιακή πολιτική, γιατί πρόκειται για ε, χρηματοδοτικού κανόνες που βασίζονται σε αποτελέσματα. Ξέρετε ότι και στη δική μας την Επιτροπή ε, αγωνιζόμαστε για περισσότερη πολιτική Όταν οι άνθρωποι υποφελούνται από κάποιους, σε κάποιους τομείς, θα πρέπει εκεί να εντείνουμε τις προσπάθειες. Αλλιώς υπάρχουν καταστάσεις, προκύπτουν καταστάσεις όπου οι άνθρωποι δεν επωφελούνται, ε, προκύπτει η διαφθορά και δεν καθίσατε δυνατό τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν σωστά. Κυρίως στον τομέα της ε, ανάπτυξης. Η απλούστευση είναι το βασικότερο. Κανονικά ε, δεν υπάρχει σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, ως εκ τούτου η λογοδοσία δεν είναι και εύκολη. Η απλούστευση νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε να έχουμε, αλλά από την μακρά μας εμπειρία γνωρίζουμε ή εγώ γνωρίζω ότι η απλούστευση τελικά δεν πρέπει να εκφυλίζεται σε υπεραπλούστευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλοι συνάδελφοι, επιθυμεί κάποιος άλλος να λάβει το λόγο, από ό,τι βλέπω όχι. Αν όχι, ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Έχουμε εκπροσώπους και από την ΤΕΦΚΟ και από την Budget. Budget, εσείς από τον προπολογισμό θέλετε να μιλήσετε πρώτος. Είσαστε από την Γενική Διεύθυνση προπολογισμού μάλιστα, Ολιβιέ Βουέλμπρουκ είναι το όνομά μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την ποιότητα της έκθεσης ε, και εμείς ε, στηρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στόχο της απλούστευσης και την ευελιξία που πολύ σωστά είπατε είναι απαραίτητα για να είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική ανάπτυξη. Ε, θα ήθελα σύντομα να σχολιάσω τις τροπολογίες σας. Ε, δεχόμαστε τις περισσότερες εξ αυτών, αλλά πρέπει να σχολιάσω τρεις. Ε, το θέμα της ευελιξίας, να σας εξηγήσουμε τι έχουμε κατά νου. Ε, να σας καθησυχάσουμε, δεν θέλουμε τα χρήματα να φεύγουν από το εργαλείο από το οποίο προέρχονται. Αυτό που επιθυμούμε είναι να υπάρχει ένα περιτόριο για να μην είναι απαραίτητο ε, να ζητάμε ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε καλύτερη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, αλλά δεν διαφωνούμε καθόλου ότι θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν κάθε ένα από τα εργαλεία από τα οποία φεύγουν αυτά τα κονδύλια. Επίσης, ε, θα θέλαμε να ενημερώνεται και το Κοινοβούλιο για τη χρήση του περιθωρίου. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι για τα καταπιστεύματα. Έχουμε συμφωνήσει ε, ως προς τον προπολογισμό του 2017. Εκεί διαπιστώσαμε ότι όσον αφορά το καταπίστευμα για την Τουρκία θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές, οι κανόνες και αναλαμβάνουν όλα αυτά να ενταχθούν μέσα στην αναθεώρηση του κανισμού έτσι ώστε να υπάρχει ε, σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και τη λογοδοσία. Ξέρετε ότι έχουμε δεσμευτεί να ενημερώνουμε τη Δημοσιονομική Αρχή να παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασίας και εκεί να φαίνεται η ε, σωστή ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Επίτροπός μας έχει προτείνει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, προτείνουν εκπροσώπους ε, στα διοικητικά συμβούλια των καταπιστευμάτων. Άρα εργαζόμεθα προς την ίδια κατεύθυνση. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωσή μας να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για το τι ακριβώς διαδραματίζεται στα καταπιστεύματα και έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε ε, σε διαρκή βάση. Εμείς προτείνουμε πρώτα να ζητείτε η γνώμη σας πριν από τη σύσταση των καταπιστευμάτων, μετά ε, να συμμετέχετε στα διοικητικά συμβούλια και επίσης ε, προτείνουμε και την ε, πιο συχνή και πυκνή ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ετήσια ενημέρωση θα παραμείνει ως έχει, θα είναι πολύ πιο λεπτομερής και εκεί θα αναφέρεται και η προστιθέμενη αξία των καταπιστευμάτων. Νομίζω ότι έχουμε προτείνει μια σφαιρική απάντηση στις ανησυχίες του ε, Κοινοβουλίου. Αυτό που δεν στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό που προτείνεται για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης για μη επίγοντα καταπιστεύματα. Σίγουρα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επίγουσα και την μη κατεπίγουσα χρήση, αλλά όπως πως ξέρετε, ε, τα καταπιστέματα ε, καλύπτουν οριζόντιες ανάγκες. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Αλλά κατά τα άλλα θέλω να πω ότι ε, πράγματι και εμείς συμφωνούμε με αυτά που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελικά όσον αφορά το περίφημο 7% Θέλω να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι αυτό ήδη εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα γνωρίζετε ότι και εμείς ε, έχουμε ορίσει το ίδιο μέγιστο ποσοστό, αλλά εδώ εσείς προτείνετε να προσθεθεί αυτό σε ένα άνθρωπο που αντιμετωπίζει πάρα πολλές καταστάσεις από τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για την περίπτωση έφταση κρατών ε, μέχρι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, και σε μελέτες ε, που απαιτούν επαΐοντες. Άρα δηλαδή αυτό το 7% καλύπτει πάρα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να αναφέρετε έναν ανώτατο όριο. Και μην ξεχνάτε ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αυξηθούν και οι δαπάνες συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους. Τις περισσότερες φορές είμαστε κάτω από 7%. Υπάρχει μια τάση να ε, διεκδικούν το ανώτατο. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερα ε, να υπάρξει μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προφανώς με αναφορά σε εσάς. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε για την απλούστευση και την ευελιξία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έμπλ. Ο κύριος. Με συγχωρείτε, ως προς τα ονόματα δεν τα πάμε και πολύ καλά σήμερα το πρωί ήμασταν σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών και λάβαμε υπόψη τα δεδομένα από αυτή τη Γενική Διεύθυνση και τα εντάξαμε στο πρόγραμμά μας. Ένα επιπρόσθετο σχόλιο στις παρατηρήσεις σας σε σχέση με την χρηματοδότηση με βάση τα αποτελέσματα σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως ε, την ανάπτυξη θα λάβουμε υπόψη τα δεδομένα ε, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορέσαμε να ε, εφαρμόσουμε τα δεδομένα εξαιτίας έκρηθμης κατάστασης και το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων ως προς τα ευρωπαϊκά καταπιστεύματα ε, αναρωτιόμαστε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτή η διάκριση μεταξύ κατεπίγουσας και post-emergency αντιμετώπισης ως προς τις κατεξιοδότηση πράξεις. και να δούμε τι γίνεται με τα καταπιστεύματα που αντιμετωπίζουν ε, έκτακτες καταστάσεις έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο πρέπει να διαλυθούν αυτά τα καταπιστεύματα και να δημιουργηθούν άλλα με βάση της κατεξιοδότηση πράξης. Ευχαριστώ. Σαλπιότ από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, με βάση τη δική μας Γενική Διεύθυνση ΕΚΟΝ συμφωνούμε απόλυτα με την ε, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας και πώς πρέπει να δράσουν ε, οι φορείς αυτοί. Αυτή η προσέγγιση της εστίασης στην προσοχή στα αποτελέσματα, focus on results, ε, δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα κυρωτικό σύστημα. Υπάρχει ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνήσει η Κομισιόν ως προς τα καταπιστεύματα βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η τάση να δημιουργούνται νέα καταπιστεύματα και δεν έγινε διαβούλευση πριν συσταθούν αυτά τα καταπιστεύματα και δεν βλέπουμε πως ε, θα γίνει αυτή η διαβούλευση και στο μέλλον. Ούτε καν μας ε, ενημερώσατε για τη σύστασή τους. Άρα δεν υπάρχει σωστός μηχανισμός, ε, ελεγκτικός μηχανισμός. Δηλαδή βγάζετε χρήματα από τον προϋπολογισμό και τα βάζετε σε μικρά δοχεία, ας πούμε, που είναι πιο ευέλικτα. Αυτό όμως μας απασχολεί. Γιατί αυτή τη στιγμή κάθε φορά που υπάρχει μία διεθνής διάσκεψη δημιουργούμε και ένα νέο καταπίστευμα. Πού θα σταματήσει αυτό. Η Επιτροπή σκέφτεται ποσοστιαίες αναλογίες για σύσταση καταπιστευμάτων. Πώς θα σταματήσουμε να δημιουργούνται αυτά τα καταπιστεύματα, να εμφανίζονται σαν μανιτάρια. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό αφορά και την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Για τη δημιουργία δηλαδή καταπιστευμάτων με κατεξουδότηση πράξης. εάν ε, δεν αφορούν βραχυχρόνια δράση, τότε θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τις ε, επί του προϋπολογισμού αρχές. Η Μαρία. Μπορώ να μιλήσω γερμανικά. Βάλτε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας θα ήθελα να στηρίξω και να υπογραμμίσω αυτά που είπε η Λίντα. Δηλαδή, πράγματι ανησυχούμε με όλα αυτά τα καταπιστεύματα, στο τέλος θα χάσουμε και τον έλεγχο. Ε, και δεν θα έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση τα λείπει από την ε, ε, ανάπτυξη εκεί που πραγματικά είναι απαραίτητο να ε, αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Αυτό ανησυχεί και έχει θορυβήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω όμως το λόγο στη συνάδελφα μου, η οποία ασχολείται με το θέμα περισσότερο από ό,τι εγώ. Ευχαριστώ. Θυμάμαι όταν αρχίσαμε να μιλάμε για την ανάγκη ευελιξίας του δημοσιονομικού κανονισμού έγινε μία συζήτηση με την Αντιπρόεδρο Γεωργίεβα στην Κωνσταντινούπολη όταν ήμασταν στη διάσκεψη ε, για τις ανθρωπιστικές ανάγκες και μας είπε ότι ολόκληρο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δεσμευτεί ως προς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαφορετικά θα υπάρχει λιγότερη ευελιξία για αυτούς που χρησιμοποιούν τα κονδύλια αυτά. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε η έλεγχη να μην είναι άκρος γραφειοκρατική. Και τώρα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολισμού θέλει συνεχείς ελέγχους. Ε, έτσι ώστε να υπάρχει μία ε, διασταύρωση δεδομένων για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βασιστεί η Επιτροπή στις ε, αξιολογήσεις. Αυτό έχει μπει στο δημοσιονομικό κανονισμό και θα πρέπει να παραμείνει, διότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θέλει επιπροσθέτους ελέγχου. Yeah. And so one question is well about the EDF money put και σε σχέση με την ε, γεωγραφικό, γεωγραφικό ε, επιμερισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, αυτά τα κονδύλια και για τις χώρες ΑΚΕ. Οκ, αυτό μου είπαν και δεν ήμουν σίγουρη. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε από πού προέρχεται το χρήμα και πού πάει. Χρειάζεται ευελιξία αλλά για τους σωστούς λόγους. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντική, λέει ο πρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών και θα πρέπει να δείτε το ότι έχουμε δημιουργήσει μόνο τέσσερα καταπιστεύματα. Ε, ε, έχουν δημιουργηθεί για τη Λιβύη, για την Κολομβία και για άλλες δύο χώρες. Για τη Μοζαμβίκια, για άλλη μία χώρα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να έχουμε μια συγκεκριμένη δράση για αυτές τις χώρες. Άρα δεν έχουμε δημιουργήσει και τόσα πολλά καταπιστεύματα. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα πλαίσια των δημοσιονομικών αρχών και την γεωγραφική κατανομή των κομβίλιων. Αυτό πώς μπορείτε να το ελέγξετε. Το ελέγχετε γιατί γίνεται ε, έλεγχος, υπάρχει reporting και μετά απαλλαγή και μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα για να έχετε πλήρη έλεγχο. Υπάρχει λογοδοσία της Επιτροπής για την διαχείριση των καταπίστευμάτων από τον ε, επικεφαλής ελέγχου, από την Όλαφ και ούτω καθεξής. Στην αρχή του άρθρου 202, 27, αναφέρουμε ότι η Επιτροπή δημιουργεί καταπιστεύματα αφού, αφού πληροφορήσει. Εγώ μπορώ να θέλω να κάνω κάτι αύριο. Ε, άλλο το να σας πληροφορήσω και άλλο να γίνει η διαβούλευση πριν λέει η πρόεδρος. Είδατε την ε, πίστολη του Επιτρόπου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνεται διαβούλευση μαζί σας και μετά να ε, διοριστούν και εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν κενά στη λογοδοσία. Όταν μεταφέρουμε κονδύλια από ένα μέσον σε έναν άλλο φορέα, τότε γίνεται ε, έλεγχος και εσείς βρισκόσαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δείτε την πραγματική εφαρμογή και σωστή και εύρυθμη λειτουργία των καταπίστευμάτων. Να ξέρετε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται και να γνωρίζετε τι ακριβώς κάνουν. Ε, γιατί και στη Λιβύη και στη Βαγδάτη υπάρχει μεγάλη κρίση και θα πρέπει να έχουμε ένα μέσο αντιμετώπισης. Επίσης θα ήθελα να σας προτείνω ε, να εγκρίνετε αυτό το μέσο ή δεν θα πρέπει να έχουμε ελέγχους επί ελέγχων όπως αναφέρεται και στο προσχέδιο της Επιτροπής Προϋπολογισμών και θα πρέπει να υπάρχει ένα πραγματικό μέσο για μείωση διοικητικού φόρτου. Για το EDF θα πρέπει να δούμε πώς έχουμε χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για κάθε γεωγραφική περιοχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Η συζήτηση λοιπόν θα συνεχιστεί και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Υπάρχει για την Ανατολική Αφρική, υπάρχει για την Κολομβία ε, ναι μεν υπάρχουν θέματα που είναι κατεπήγοντα αλλά είναι στην ουσία κάτι το οποίο έχει ξεφύγει θα έλεγα από τις κανονικές διαδικασίες προσπάθειες έβρεσης πιστώσεων. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το θέμα της έβρεσης μελών για τα διοικητικά συμβούλια των καταπίστευμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα αυτό. 28 Μαρτίου 12 12η μεσημβρινή προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Να πω ότι λόγω της ειδική ε, ολομέλειας τελετής για τα 60 χρόνια της συνθήκης έχουμε αναβάλει το 12 για τη μείωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και περνάμε στο 13 ε, για φορολογικές δηλώσεις και στοιχεία φορολογικά από ορισμένου τύπου ε, οργανώσεις και οντότητες. Έχετε πολύ λίγο χρόνο στην διάθεσή σας. So can we invite our guests, two guest speakers come sit? We have space here, maybe. Έχουμε δύο προσκεκλημένους ομιλητές, μπορούν παρακαλώ να έρθουν στο Προεδρείο. Okay, so, um, this... Καλώς λοιπόν θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων για την γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ και για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τη δημοσίευση στοιχείων φόρου εισοδήματος από συγκεκριμένες κατηγορίες εταιριών είναι τμήμα του πακέτου καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Πρόκειται επίσης για την πρωτοβουλία BETS, για την καταπολέμηση δηλαδή της μείωσης της φορολογικής βάσης, της συρρήκνωσης της φορολογικής βάσης. Να το πω αλλιώς είναι τα παραθυράκια που επιτρέπουν σε ορισμένου τύπου επιχειρήσεις να αποφεύγουν να πληρώνουν φόρους. Απαιτείται σήμερα από τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις να δημοσιεύουν στοιχεία φορολογικά εκεί όπου πληρώνουν φόρους. Εταιρείε πάνω με πάνω από 75 εκατομμύρια κύκλο εργασιών ε, θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένες και διαφανείς σε σχέση με το που δηλώνουν ε, τα φορολογικτέα τους έσοδα. Αλλά για τις μικρότερες επιχειρήσεις τα πράγματα είναι κάπως συγκεχημένα. Είχαμε την έκθεση το 2015, ε, ε, ε, την έκθεση πάλι της κυρίας Σλάιν για τις χώρες τις οποίες υπήρχαν συστήματα φοροαποφυγής. Στις αναπτυσσόμενες χώρες λένε τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι υπάρχει μια 20% διαφορά ανάμεσα στους συλλεγόμενους φόρους και στους προβλεπόμενους προσυλλογή φόρους. Συνεπώς λοιπόν έχουμε και δύο εμπειρογνώμονες από την Oxfam και την Eurodap και θα τους δώσουμε το λόγο. Η κυρία Σαρντονέ από την Oxfam. Έχετε 8 λεπτά. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε, την Oxfam δηλαδή, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, λειτουργούμε σε 90 χώρες προωθώντας την ισότητα ε, και διαπιστώσαμε εδώ και χρόνια τη μεγάλη σημασία που έχει το δίκαιο φορολογικό σύστημα και η διαφάνεια η φορολογική. Τον προηγούμενο Ιανουάριο η Oxfam δημοσίευσε μια έκθεση και αναφερθήκαμε στην εξαιρετικά υψηλή ανισότητα η οποία έχει αρχίσει δυστυχώς να αυξάνεται ακόμα περισσότερο τα τελευταία 25 χρόνια. Αναφερθήκατε εσείς στα 100 δις τα οποία χάνονται για τις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της διαφυγής ε, πληρωμής φόρου από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Όπως λοιπόν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα τα φορολογικά όπως γνωρίζετε επίσης, πολλές χώρες αποφάσισαν ότι τα στοιχεία αυτά δεν δίδονται στις υποανάπτυξη χώρες. Όταν υιοθετήθηκε στα πλαίσια των διαδικασιών του ΟΣΑ το σύστημα της έκθεσης αναχώρας, εξαιρέθηκαν οι χώρες αυτές. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τις φορολογικές υπηρεσίες που κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά ζητάμε απλά να εφαρμόζονται οι κανόνες, δεν ζητάμε να υπάρξει μια αλλαγή των κανόνων. Είναι βασικό λοιπόν να ελέγχεται αναχώρα το σύστημα έτσι ώστε να δούμε αν πράγματι υπάρχει διαφυγή στον τομέα της ίσπραξης φόρων Πολλές χώρες αναπτυσσόμενες όμως έχουν ε, ε, επιχειρήσεις πολυεθνικές με την έδρα τους στις συγκεκριμένε χώρες αλλά ελάχιστα φορολογικά έσοδα και δεν μπορούν να γνωρίζουν πού και πόσο πληρώνουν οι συγκεκριμένες αυτές ε, επιχειρήσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αρκετά στοιχεία από τον πιστοτικό τομέα. Η Oxfam Γαλλίας πέρυσι μαζί με άλλες ΜΚΟ δημοσίευσαν μία έκθεση μετά από την δημοσιοποίηση των κερδών γενικά και του κύκλου εργασιών των γαλλικών τραπεζών στο σύνολο του κόσμου ε, και επίσης ε, δηλώνουν τα κέρδη που είχαν στις αναπτυσσόμενες χώρες και τους φόρους που πληρώνουν στις συγκεκριμένες χώρες. Όταν μιλάμε για ανισότητες, εδώ βλέπετε ότι οι γαλλικές τράπεζες κερδίζουν 43.000 ευρώ ανά υπάλληλο ουσιαστικά ενώ βλέπετε ότι στις υπόλοιπες χώρες ε, το ποσοστό είναι πολύ ε, χαμηλότερο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτή η ανισότητα από πραγματικά ουσιαστικά θέματα. Την επόμενη εβδομάδα η Oxfam θα κυκλοφορήσει μια νέα έκθεση για τις 20 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και θα δείτε ότι οι ανισότητες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Θα σας στείλουμε την έκθεση αυτή για να δείτε κι εσείς πώς δουλεύουν οι τράπεζες στη δική σας χώρα. Να επανέλθω τώρα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΟΟΣΑ λοιπόν επιτρέπει και η ομάδα των 20 να κατακρατούνται ορισμένες τέτοιου είδους πληροφορίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες να είναι πιο προοδευτικές και δημοκρατικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δική της πρόταση υποχρεώνει τις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις να δηλώνουν τις δραστηριότητές τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι αναχώρα. Θεωρείται ότι αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά το θέμα είναι να δούμε τι συνέπειες έχει και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Καταρχάς ε, βρίσκονται πάντα στο σκοτάδι οι αναπτυσσόμενες χώρες και το δεύτερο που θα ήθελα να πω ε, αν έχει κανείς συγκεντρωτικά στοιχεία για συγκεκριμένες χώρες μπορεί να δει κανείς τι βγαίνει και τι μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να συγκρίνει αριθμούς ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ισπανία ή τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί κανείς να ζητήσει να αναπτυχθούν νέα προγράμματα ελέγχου αλλά δεν μπορεί να τα επιβάλλει. Ένα επιπλέον στοιχείο στα πλαίσια της πρότασης είναι ότι συνδέει την πρόταση αυτή με τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων. Αυτό ξεκίνησε μία εβδομάδα μετά από το Panama Papers ε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στους φορολογικούς παραδείσους. Ε, έγιναν λοιπόν κάποιες διευρύνσεις της εμβέλειας της ρύθμισης, αλλά ακόμα και σήμερα δεν έχει κυκλοφορήσει ε, η μαύρη λίστα, ίσως να μην υπάρχει τίποτα μέσα στη μαύρη λίστα, διότι η Προεδρία της Μάλτας στην τελευταία συνάντηση κορυφής ήταν ότι εμείς θα θέλαμε να κενώσουμε ουσιαστικά τη μαύρη λίστα, οπότε μπορεί και να μην υπάρχει πλέον. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι η μοναδική λύση για να υπάρχει μια έκθεση αναχώρα είναι να υπάρξει διαχωρισμός των στοιχείων αναχώρα ανά μεγάλη επιχείρηση. Αυτό επηρεάζει και την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα του ανταγωνισμού. Και δεν είναι κάτι που θίγει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ε, θα πρέπει λοιπόν τα στοιχεία που θα προκριθούν να είναι χρήσιμα και για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους πολίτες ε, από τρίτες χώρες. Τεμέγερ. Thank you very much, and thank you for your kind invitation to present on public country by country reporting in front of the Development Committee. Uh, My name is Το όνομά μου είναι Ντεμέ και εγώ εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανάπτυξης και ασχολούμαι με θέματα φορολογικής δικαιοσύνης. Ε, η έκθεση αναχώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Eurodac και άλλοι ε, έχουν ζητήσει από το Φεβρουάριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ε, τον Απρίλιο του 2016 με χαρά ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε νομοθετική πρόταση έτσι ώστε να δημοσιοποιείται, δημοσιοποιούνται οι εκθέσεις αναχώρα. Εμείς το είχαμε ζητήσει όπως ξέρετε πριν από αρκετά χρόνια. Πάντα Πάντως ε, σύντομα γρήγορα απογοητευτήκαμε και ακούσαμε ότι η πρόταση Κομισιόν θα καλύπτει μόνο τις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και κάποιους φορολογικούς παραδείσους. Θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Για λόγους που έχει πει η Oxfam, αυτό είναι ένα κενό μέσα στο κείμενο της οδηγίας. Εγώ στην παρέμβαση μου θέλω να εστιάσω σε κάποια άλλα στοιχεία που λείπουν από την πρόταση της Επιτροπής. Πρώτον, όσον αφορά το κατόφλι της ε, αναφοράς. Ξέρετε ότι το κείμενο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ότι οι πολυεθνικές με 750 εκατομμύρια ευρώ τζίρο ε, αυτές θα κληθούν να αναφέρουν αναχώρα. Με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ αυτό το κατόφλι σημαίνει ότι το 85 μέχρι 90% των πολυεθνικών δεν θα χρειάζεται να λογοδοτούν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει ότι πολλές πολυεθνικές θα αποκλειστούν από τη λογοδοσία αναχώρα ε, το στοιχείο, αυτό το κατόφλι είναι πολύ προβληματικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές είναι κάτω από 750 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών και επίσης αυτές οι αναπτυσσόμενες ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του το έχουν από εταιρικούς ε, φόρους. Άρα δηλαδή εδώ θα εμπίπτουν οι πολύ μικρές εταιρείε. Παράδειγμα, στη Σιέρα Λεόνε το 2013 οι εταιρείε εξόριξης Σιέρα, Ρατάιλ και Μάντα Μάινινγκ είχαν το 3% και το 10% του ΑΕΠ της χώρας, τη Σιέρα Λεόν. Αυτό προσπορίστηκαν. Κάτω δηλαδή από τα 750 ε, εκατομμύρια ευρώ. Και από εκείνο όμω πάνω που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να γίνει ε, λογοδοσία στη Σιέρα Λεόν. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος ορισμός ε, για τη λογοδοσία σε άλλα στοιχεία από τα ποσά που αναφέρονται στο τζίρο. 40 εκατομμύρια παραδείγματο χάρη. Ναι. Αυτό το ενέκρινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, ε, ασχολήθηκε με την οδηγία περί των δικαιωμάτων μετόχων ε, που ψηφίστηκε το 2015. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο λείπει από την πρόταση της Επιτροπής είναι ότι δέχεται ότι λείπουν σημαντικά στοιχεία ε, που δεν κοινοποιούνται, Παραδείγματο χάρη με βάση την πρόταση της Επιτροπής, οι πολυεθνικές ε, δεν είναι υποχρεωμένες να αναφέρονται στις αγορές και τις πωλήσει σε κάθε χώρα, ε, στην αξία των ε, ενεργητικών στοιχείων ε, της ε, εταιρεία σε κάθε χώρα. Λείπουν και κάποια άλλα στοιχεία που δεν χρειάζεται να αναφέρονται οι εταιρείε. Νομίζω αυτά περιλαμβάνονται και σε αυτή την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των μετοχών. Επειδή λοιπόν δεν θα υπάρχουν στοιχεία για τα κεφάλαια και τις δραστηριότητες των πολυεθνικών θα είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες ε, να μπορέσουν να έχουν μια εικόνα για το τι κάνουν οι πολυεθνικές στη χώρα τους. Δηλαδή ε, η κοινή γνώμη ε, θα έχει περιορισμένη πληροφόρηση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται περισσότερα στοιχεία για να γνωρίζει κανείς καλύτερα που ακριβώς διεξάγουν τις δουλειές τους οι πολυεθνικές και έτσι να είναι δυνατόν να υπάρχει και καλύτερη αξιολόγηση ποιοι φόροι καταβάλλονται σε κάθε χώρα. Αυτό με βάση την αρχή ότι οι πολυεθνικές πρέπει να καταβάλουν φόρους εκεί που κάνουν δουλειές και εκεί όπου αποκομίζουν ωφέλη από τις κοινωνίες και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, απαιτεί μόνο από τις πολυεθνικές, ε, να, μάλλον ζητάει από τις πολυεθνικές να δημοσιεύουν αυτά τα στοιχεία μόνο στις ιστοσελίδες τους. Άρα δηλαδή όποιος θέλει να αναλύσει πληροφορίες πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα της ε, πολυεθνικής μόνος του να μπαίνει κανείς σε, κάθε ιστοσελίδα για να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πολύ επίπονη δραστηριότητα που περιορίζει τη δυνατότητα των κοινωνιών των πολιτών να αναλύουν τις πληροφορίες. Η ε, Κομισιόν δεν αναφέρει ποιο είναι ε, το, ποιο, είναι το πρότυπο εκείνο ε, που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ε, και με τον τρόπο αυτό ε, δεν μπορεί να γίνει και σύγκριση. Επίσης, πολύ πιο λογικό θα ήταν να απαιτηθεί οι πληροφορίες να παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο πρότυπο και έτσι οι κοινωνίες των πολιτών να μπορούν να αναλύουν τις πληροφορίες. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η αναφορά αναχώρα θα πρέπει να καλύπτει όλες τις χώρες, το κατόφλι αναφοράς να είναι χαμηλό, να αποκαλύπτονται πολλά στοιχεία και να δημοσιοποιούνται όλα αυτά σε ένα εύκολα προσπελάσιμο μητρό. Ε, να είναι κοινό το πρότυπο. Αυτά όλα είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η νομοθεσία έχει νόημα, βοηθάει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να μην υπάρχει ε, αποφυγή, φοροαποφυγή εταιρικών φόρων να μην βρίσκονται ε, επίση ε, αναπτυσσόμενες χώρες στο σκοτάδι, δηλαδή να μην μπορεί κανείς να μάθει τίποτα για αυτές. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και με μεγάλη μου χαρά να δεχτώ ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μήπως μπορείτε και να κλείσετε και το μικρόφωνο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, έχουμε τη γνωμοδότηση της κυρία Σλάιν και τώρα Έλλη ε, θα ήθελα να σου δώσω το λόγο για να απαντήσεις. Ευχαριστώ Λίντα και ευχαριστώ την Oxfam και τη Eurodat για την παρουσίασή τους. Τα έγγραφα του Παναμά δείχνουν ότι είναι παγκόσμιο το θέμα και χρειάζονται και παγκόσμιες λύσεις. και θεωρώ ότι οι μεμονωμένες προσπάθειες είναι καταδικασμένες. Μιλήσαμε λοιπόν για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων από πλευράς αναπτυξιακής πορείας και ως προς που καταβάλουν το υψηλότερο τμήμα. Τίμημα, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν τις ε, πιο απλές υπηρεσίες με το πιο απλό τρόπο. Θεωρώ ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τα έσοδά τους για την ανάπτυξη κατά 20%. Αυτό μπορεί να γίνει με τη δίκαιη φορολόγηση. Ορισμένα από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ καλά βήματα, αλλά δεν χρησιμεύουν στον υποανάπτυξη κόσμο. Όπως ελέγχθη, ε, αυτή η πρόταση μένει πολύ πίσω για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των πολυεθνικών που μπορούν να φοραποφύγουν σε φτωχές χώρες, γιατί υπάρχει κάλυψη των ε, πολυεθνικών και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση αναχώρα αλλά θεωρώ ότι η πρόταση δεν είναι σωστή και είναι άχρηστη για τις υποανάπτυξη χώρες γιατί δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε πλήρη αποτίμηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την εκμετάλλευση των ε, αναδυόμενων οικονομιών και των υποανάπτυξη χωρών. Με βάση την πρόταση του 2015 θα πρέπει να ε, αποκαλύπτουν τα στοιχεία σε όλες τις χώρες της ε, Αφρικές. Όμως η πρόταση αυτή οδηγεί σε φοροαποφυγή και δεν προβάλλει την ανάπτυξη. Δεν μιλάμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αναπτυσσόμενες χώρες χάνουν δισεκατομμύρια ετησίως. Θα πρέπει λοιπόν να μην παίρνουμε με το ένα χέρι αυτό που δίνουμε με το άλλο. Η πρόταση γνωμοδότηση προς την ΕΚΟΝ προσπαθεί να διορθώσει αυτά τα μεγάλα χάσματα στην πρόταση της Επίτροπης. Θα θέλαμε στοιχεία ε, όχι σε συνολικό επίπεδο και ένα κατώτερο κατόφλι, γι' αυτό ζήτησα να λάβουμε υπόψη τις μεγάλες ε, ε, επιχειρήσεις με κατόφλι 14 ε, εκατομμύρια. Μόνο με μια μεγάλη δέσμευση αντιμετώπισης της φοροαποφυγής θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παγκοσμίως. Θα θέλαμε λοιπόν να δίδονται περισσότερα στοιχεία σε, ε, σε μία μορφή με κοινά πρότυπα. Πιστεύω ότι έτσι θα φτάσουμε στα πιο φιλόδοξα αποτελέσματα. Σκιώδης. Τώρα ο κύριος Ρούμπιχ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά ε, κυρίως ε, την Oxfam για την εισήγησή της, διότι η διαφάνεια κυρίως ε, σε θέματα φορολογίας είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν έτσι μια καλή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τα χρήματά τους. Και ειδικά στην ε, αναπτυξιακή πολιτική είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι δηλαδή οι αρμοδιότητες προβλέπονται μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 και βεβαίως για περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα είναι ένα θέμα. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Πάντως εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά τις ε, προϋποθέσεις για την χορήγηση βοήθειας και ενισχύσεων, πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Να ξέρουμε πώς ε, χρησιμοποιούν τα χρήματα η ΜΚΟ, παραδείγματος χάρη, ή οι δημόσιοι οργανισμοί. Και ε, με, αυτούς τους, ε, με αυτές τις εκθέσεις αναχώρα είναι επίσης σημαντικό να βλέπουμε κατά πόσον τα χρήματα παραμένουν εκεί όπου προκύπτει τη προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αρχή και πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε πού προκύπτουν τα κέρδη, οι ε, μεγάλες εταιρείες ε, κατά κάποιον τρόπο προστατεύονται προστατεύονται από την παρέμβαση ε, των ε, εφοριακών αρχών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυστυχώ αναγκασμένες να τα αποκαλύπτουν όλα με απόλυτη διαφάνεια και με λεπτομέρειες. Η διαφάνεια λοιπόν στις ε, μεγάλες εταιρείες θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση καταβολής φόρων μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. Εμείς επιθυμούμε κυρίως οι οικογενειακές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες να έρθουν σε επαφή με οικογενειακές επιχειρήσεις εδώ στην Ευρώπη. Και με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορούσε να προκύψει μια φορολογίας για ε, επιτιδευματίες, για γυναίκες, ε, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ελκυστικότητα να αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανεί σε όλου αυτού του τομεί. Και για τι μεγάλε εταιρείε είναι σαφέ ότι έγιναν μεγάλε γιατί εκμεταλλεύτηκαν μονόπλευρα και μονομερό ωφέλη. Ε, γνωρίζουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φόρων που καταβάλλονται στην Ευρώπη είναι από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και από τους εργαζόμενους τους. Οι μεγάλες φορολογούνται κατά κανόνα, μόνο το 4% φορολογούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει λοιπόν κάποια ισορροπία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό καθήκον ε, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε όλοι μας. Ε, ως εκ τούτου για μένα αυτή, αυτές οι εκθέσεις αναχώρα πραγματικά είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ Γκέρνς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν βλέπω γιατί να εφαρμόσουμε τα ανώτατα όρια μια επιχείρηση. Δεν είναι καλή όταν είναι μικρή και δεν είναι κακή υποχρεωτικά όταν είναι μεγάλη, πάνω από 750 εκατομμύρια. Αυτός ο δετερμινισμός νομίζω με βάση τον κύκλο των εργασιών είναι λάθος ανεξαρτήτως του ύψους των κερδών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και εδώ θα κάνω μια δεύτερη παρατήρηση. Αν εφαρμόσουμε τα όρια θα υπάρχουν πάντα παραθυράκια έτσι ώστε να μην υπόκεινται στην διαφάνεια που απαιτείται κάποιες επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιούν κάποιες επιχειρήσεις με μικρότερο κύκλο εργασιών κτλ. Θεωρώ επίσης ότι είναι και λίγο πατερναλιστική η αντιμετώπιση. Εμείς είμαστε αυτοί που θα επιβάλλουμε και θα ορίσουμε τον νόμο. Ε, εντάξει, αλλά αυτό έχει σχέση και με τα κοινοβούλια των συγκεκριμένων χωρών, οι οποίες θίγονται από την μη καταβολή των φόρων, πόσο μάλλον που μετά από την θέση σε ισχύ των εταιρικών συμφωνιών υπάρχει ένας φορολογικό έσοδο το οποίο θα εξαφανιστεί. Ξέρουμε ότι η φόροι εισαγωγή, σαν παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες ε, υπό ανάπτυξη θα πρέπει να αντικατασταθούν από κάποιους άλλους ε, πόρους έτσι ώστε να καλύπτονται οι οικονομικές ανάγκες. Ναι μεν λοιπόν υπέρ της διαφάνειας φυσικά, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα και η διακυβέρνηση των χωρών εταίρων να είναι τέτοια έτσι ώστε τα παραθυράκια να είναι κλειστά και μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης ε, να κάνουμε τα απαραίτητα. Αυτά για τις χώρες οι οποίες ε, θα έλεγα έχουν έσοδα από αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις εκθέσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου για τα θετικά στοιχεία της πολιτικής μας μέχρι τώρα στον τομέα αυτό. Μια ερώτηση να κάνω τώρα προς τους δύο εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Τι γίνεται ε, με την ρύθμιση Dodd Frank στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρύθμιση αυτή η νομοθετική μπορεί να μετριάσει την έλλειψη διαφάνειας οι χώρες οι οποίες επιβάλλουν την καθολική επιβολή φόρου όπως τις Ηνωμένε Πολιτείες ενός τύπου διαχειρίζονται τα προβλήματα αυτά καλύτερα, προλαμβάνουν καλύτερα την διαφυγή φόρων. Ε, παράδειγμα στην Ελλάδα. Ε, λέμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιβάλλει φόρους στους πλούσιους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό όταν είστε πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είτε ζείτε στην Ναμίμπια, στην Νότιο Αφρική, στο Βέλγιο ή στη Γερμανία, πληρώνετε φόρο στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Νομίζω λοιπόν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, και μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το οποίο λέγω, νομίζω ότι και αυτό θα ήταν μια κάποια λύση. Ναι, ναι στην διαφάνεια, έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα διαφάνειας εθελοντικής στα πλαίσια του Global Compact που ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τίποτα να κρύψουν και συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, αλλά τελικά θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν και θα πρέπει η πολιτική μας δράση να μπορέσει να δώσει αποτελέσματα αυτά. Σάντσες. Ευχαριστώ. Όπως έγινε πρόσφατα στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο με τη Fiat και ε, τη Starbucks ή με την περίπτωση InBev στο Βέλγιο, Υπάρχουν και αντίστοιχες τέτοιες καταστάσεις και στην Ιρλανδία. Θεωρείται ότι στην ουσία οι διευκολύνσεις οι φορολογικές αυτές είναι παράνομες επιδοτήσεις. Θα πρέπει να τεθεί τροχοπέδι στην εκροή φορολογικών εσόδων. Νομίζω ότι αν δεν είμαστε αυστηροί δεν θα το πετύχουμε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει όλες τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σκάνδαλο της Apple ε, δείχνει ότι ελείπει η εγγύηση, θα έλεγα, ε, καταπολέμησης των παράνομων πρακτικών. Νομίζω ότι η Apple είναι παράδειγμα πολλών τέτοιων πανίσχυρων εταιριών που έχουν επανειλημμένα καταγγελθεί για παράνομες πρακτικές οι οποίες διαφεύγουν του σωστού δημοσίου ελέγχου. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, σε ένα πλαίσιο φιλελευθεροποίησης και λιτότητας απαράδεκτο να τα πληρώνουν όλα η μεσαία τάξη και οι εργαζόμενοι, ενώ οι πολιεθνικές να μην συνεισφέρουν ανάλογα ε, στις δομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εγγυηθούν τα υψηλά τους έσοδα. Τελειώνοντας να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έσοδα από επιχειρήσεις έπεσαν 28% ανάμεσα στο 2006 και το 2004 από 1,2 του ΑΕΠ σε 1,5 ενώ τα έσοδα βέβαια των επιχειρήσεων αυξήθηκαν και σε επίπεδο ΦΠΑ υπήρξε αύξηση και σε επίπεδο κοινωνικών συνεισφορών. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται γιατί από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ισχύσει αυτό και για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 750 ε, εκατομμυρίων. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία ε, είναι προβληματική ιδιαίτερα όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και για τις υποανάπτυξη χώρες και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, με κύκλο εργασιών κάτω των 750 εκατομμυρίων που είναι οι βασικοί επενδυτές στις χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Τα ποσά αυτά στην ουσία είναι στο ίδιο επίπεδο με τα ετήσια έσοδα τα, της, του Μπουρούντι και της Λιβερίας έχει νόημα το 750 εκατομμύρια μόνο αν θέλουμε μια οδηγία εντελώς συμβολική χωρίς πρακτικά αποτελέσματα. Να είμαστε σαφείς ότι κατά τη διάρκεια εμείς αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου δεν έχουμε δείξει την απαιτούμενη ε, επιμονή για την καταπολέμηση της φορολογικής διαφυγής. Ε, φοροδιαφυγής μάλλον και ευχαριστώ ανθρώπους όπως η κυρία Σαρντονέ και βέβαια είναι το θέμα ότι η επιδίωξη ίσπραξης των φόρων δεν θα πρέπει να θέσει σε αμφισβήτηση την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως το προβλέπουν και τα κοινοτικά μέτρα και το BEPS του ΟΣΑ. Τελικά, η έκθεση αναχώρα, δημοσιοποιημένη έκθεση αναχώρα, θα βελτιώσει τον έλεγχο των επιχειρήσεων και θα επιτρέψει στους νομοθέτες, ε, τα νομοθετικά σώματα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μόνο αν γνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους διαφεύγουν το φόρο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό αυτό. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι όλοι γνωρίζουμε ότι στην ουσία ε, η εξουσία επιδιώκεται να καλυφθεί από μια ελίτ ε, επιχειρηματικών συμφερόντων που επιβάλλει τη λιτότητα και καλλιεργεί τον λαϊκισμό και την ευρωφοβία. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για την εργασία της Ellis Line στο σχέδιο αυτό. Τα τρία βασικά σημεία είναι να έχουμε συνολικά στοιχεία από όλες τις τρίτες χώρες όπου λειτουργούν πολυεθνικές και χαμηλότερο κατόφλι για reporting 40 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης ε, μιλά για δημόσια μητρώα, καταχώρησης και για όλα τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Θα θέλαμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ποιότητα, αλλά όλα αυτά δεν ε, πρέπει να είναι μόνο ευσεβείς πόθη. Τα καταφέραμε πολύ καλά γιατί ξεκινήσαμε από την οδηγία των μετόχων που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και περιελάμβανε αυτή την ε, τροπολογία για υποβολή εκθέσεων αναχώρα με μια πολύ μικρή πλειοψηφία και στην Επιτροπή Γιούρη και στην Ολομέλεια. Όμως η Επιτροπή μας έδωσε μια οριζόντια πρόταση, γι' αυτό νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η εργασία μας. Δεν ξέρω αν άλλοι συνάδελφοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Θα ήθελα να, να πω κι εγώ ε, λίγα πράγματα. Νομίζω ότι ακούσατε για την έλλειψη φιλοδοξίας από πλευράς της ε, Επιτροπής. Ε, μετά το 2008 θεωρήσαμε ότι δεν μάθαμε, δεν διδαχτήκαμε από το μάθημα της ύφεσης του 30 και έχουν περάσει τόσα χρόνια, εννιά χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης και τώρα ίσως και στη ΣΥΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ορισμένες συστάσεις του όσα υπάρχει απεσιοδοξία σε σχέση με το κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε την φορολογική κατάσταση. DG Σίσμα και μετά Ντεύκο η Μαρία Μοντέρο ε, η Γενική Διεύθυνση Σίσμα έχω τα σωστά ονόματα ο κύριος Ραμπή έχει το λόγο εκτός μικροφώνου Δεν είσαστε τακτικό στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, κοιτάξτε κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μάλλον ε, πρόκειται για ένα ε, ακρονίμιο αυτό το οποίο σας ανέλησα, το οποίο όμως δεν αντικατοπτρίζει οπωσδήποτε αυτό το οποίο κάνουμε. Να επανέλθω στο θέμα μας. Η φύσμα είναι αρμόδια για αυτή την πρόταση και όχι η ταξούντ. Γιατί υποτίθεται εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα διαφάνειας. Και δεν έχουμε να κάνουμε με ένα καθαρά ε, χρηματοδοτικό εργαλείο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει και μια διάσταση απόψεων ανάμεσα σε εκείνους που τοποθετούν τόσο πολλές ελπίδες σε αυτό το εργαλείο, αφενός και αφετέρου ε, στο στόχο που έχει η Γενική Διεύθυνση Φύσμα ε, και αυτή η πρόταση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να αυξηθεί η ζήτηση για διαφάνεια και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο του αγώνα κατά ε, της φοροδιαφυγής. Όμως αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό όσο άλλα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν κάτω από την προοπτική της γενικότερης ε, δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Και αυτό είναι μια πολιτική προτεραιότητα για αυτήν την Επιτροπή. Επίσης, όσον αφορά στην έλλειψη φιλοδοξιών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει λιγάκι να το υποβαθμίσουμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρώτη η οποία προτείνει αυτό το συγκεκριμένο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν η μόνη που θα ζητούσε με βάση νομοθεσία ε, τη διαφάνεια. Δεν υπάρχει νομολογία επ' αυτού του θέματος. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στο θέμα της διαφάνειας. Τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η Επιτροπή να δούμε τι εγκρίθηκε πέρυσι. Αναφέρομαι στην οδηγία για την διοικητική συνεργασία. Εκεί οι αναφορές αναχώρα ε, κρίνονται υποχρεωτικές ε, από τις πολυεθνικές ε, να υποβάλλονται δηλαδή τα στοιχεία των πολυεθνικών στις φορολογικές αρχές και να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση, ε, και λόγω του ότι προβλέπεται να υπογραφεί μία σύμβαση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω τώρα ακριβώς κατά νου τα στοιχεία, αλλά ε, υπάρχουν περίπου 30 νομοθετικές αποφάσεις που καθιστούν ομολογία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιαπωνία, Κίνα, και πολλές άλλες ε, νομοθετικές αποφάσεις. Η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με φορολογικές αρχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική ε, και υπάρχουν χώρες που έχουν υπογράψει και από τις οποίες οι φορολογικές αρχές ε, θα παίρνουν πληροφορίες που σημαίνει ότι θα παίρνουν πληροφορίες ε, από πολυεθνικές. Κατ' ουσία λοιπόν τι χάνουμε. Με την πρότασή μας είμαστε επίκαιροι. Και υπάρχουν στοιχεία αναλογικότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κάναμε μία ενδελεχή ανάλυση επιπτώσεων. Ξετάσαμε το να υπάρχει ε, χαμηλότερο όριο, κατώτατο όριο, όλα αυτά δηλαδή τα οποία συζητήσαμε σήμερα. η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως να μην σας φαίνεται τόσο φιλόδοξη όσο τα έπρεπε. Και αυτό κυρίως για λόγους αναλογικότητας. Παραδείγματο χάρη, όταν λέμε ότι το ε, κατώτατο όριο είναι πολύ υψηλό, αυτό καλύπτει περίπου 6.000 ε, πολυεθνικές και αυτό περιλαμβάνει περίπου 10 μέχρι 15% των ε, πολυεθνικών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, την ίδια στιγμή καλύπτει και το 90% των ε, δραστηριοτήτων των πολυεθνικών. κατεβάζοντας το όριο από τα 750 εκατομμύρια σε χαμηλότερο επίπεδο, Αυτό σημαίνει ότι πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ε, εταιριών που θα καλούνται να καταβάλουν δηλώσεις με τον ε, ε, πολλαπλασιαστή του 10. Άρα δηλαδή Θέλουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αναλογικότητα. Και λόγος είναι γιατί η Κομισιόν κάνει αυτή την πρόταση. Διότι σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλες προτάσεις που αφορούν σε εκθέσεις αναχώρα και έχουν ήδη κατατεθεί. Σε αντίθεση λοιπόν με όλε τι προηγούμενε, αυτή η πρόταση της Επιτροπής έχει κατά νου να καλύπτονται και πολιεθνικέ εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης, που σημαίνει πολιεθνικέ οι οποίε ε, είναι εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή όμως αναπτύσσουν δραστηριότητε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς προτείνουμε να καλύπτονται και αυτέ από την οδηγία και να καταθέτουν ε, την έκθεσή τους αναχώρα όπως ακριβώς προβλέπεται. Βεβαίω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μία σειρά πληροφοριών ε, από αυτές τις εταιρείε, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και το τι είναι λογικό. Διότι δεν πρόκειται μόνο για τους φόρους που έχουν, αν έχουν καταβάλει, πρόκειται και για μία σειρά άλλων πληροφοριών που ε, προβλέπει αυτή η έκθεση. Ας πούμε, πληροφορίες για τον αριθμό των υπαλλήλων, ε, για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, για τα κέρδη Ως εκ τούτου, σας είπα, πρέπει να υπάρχει μία αναλογικότητα σε αυτά τα οποία ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις ε, εταιρείε. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν η κριτική που σας ασκείται ότι αυτή η πρόταση δεν προβλέπει το να δίδονται ικανοποιητικέ πληροφορίε για το τι συμβαίνει σε όλε αυτέ τι χώρε. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κριτική, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσαμε η έκθεση να προσφέρει τι σημαντικέ πληροφορίε. Υπάρχει ένας κατάλογος ε, χωρών όπου δεν, υπάρχει, δεν έχουμε σωστή διαχείριση. Και αν ε, προκύπτει κάποια διασύνδεση ανάμεσα σε φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με φορείς αυτών των ε, εταιριών ή των χωρών, εμείς προτείνουμε να αποκαλύπτονται πλήρως τα στοιχεία λειτουργίας των χωρών ή των εταιριών. Με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν αντιμετωπίζει τους κινδύνους και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Ε, με συγχωρείτε, 11.30 τελειώνουμε. Έχουμε την ε, εορταστική εκδήλωση. Η ώρα είναι ε, περίπου και 25. Ε, αν έχετε καλοσύνη να συντομεύετε. Με συγχωρείτε πολύ που σας διακόψα, αλλά ξέρετε, είναι η 60η επέτειος και εμείς θέλουμε να πάμε. Ε, λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, κοιτάξτε, ε, το ότι ε, ως Επιτροπή δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση και Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία της πρότασης, για μας ε, η λέξη κλειδί είναι η αναλογικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ζητώ συγγνώμη που ε, σας είπα ότι πρέπει να μιλήσετε έτσι εντάχει. Η Ντεύκο έχει κάτι να μας πει, πολύ γρήγορα όμως. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Φίσμα και υποστηρίζουμε την ε, παρουσίαση της πρότασης. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερος τρόπος να υπάρχουν ε, θελούσιοι μηχανισμοί σε διάφορα επίπεδα. Στην ΤΕΦΚΟ λοιπόν, Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, προσπαθούμε να δώσουμε τα μέσα στις χώρες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα μέσα στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και σε διμερές επίπεδο κινούμαστε και σε περιφερειακό έτσι ώστε να έχουμε South-to-South -south cooperation και προσπαθούμε να ε, καταστήσουμε αυτοδύναμες τις περιφερειακές αρχές. Έτσι ώστε να δούμε και το Ταντάτ τι καταφέρνει επιτοπίως. Ε, όπως ξέρετε η Επιτροπή συγκρότησε αυτό το μέσο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό μεταξύ άλλων, άλλων προσπαθειών μέσα στα πλαίσια του EITI. Ίσως αργότερα μπορούμε να δούμε το θέμα αυτό το, της φορολόγησης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Διαφωνούμε ως προσορισμένα στοιχεία, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αυτό το μέσον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις παγκόσμιες ανισότητες. Αυτό είναι το μέλημά μας. Εάν λάβουμε υπόψη την πολιτική συνοχής για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό θα είναι ύψη της σημασίας, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν τα ίδια μέσα για να χρησιμοποιήσουν την φόρο αποφυγή και φόρο διαφυγή των μεγάλων επιχείρησεων. θα μπορούσαμε να λάβουμε ε, υπόψη ότι ε, τελικά όλα τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι τις ε, μεγάλες φοροαποφυγές. Ωραία. Την Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 12 είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στην Επίτροπη πίστις στις 25 Απριλίου. Στις 3 η ώρα εδώ θα μιλήσουμε για ένα ειδικό θέμα. Και θα ήθελα να πω ότι ο Τσίστον είναι εδώ για τελευταία φορά και θα ήθελα να τον ευχαριστήσουμε για την εργασία του τα τελευταία χρόνια.